διαχείριση εμπορευμάτων καταγωγή η σημερινού και δίνω το λόγο για τέσσερα λεπτά στον εισηγητή. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση έχει σημαντική προϊστορία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο παρελθόν συνήψαν δύο σημαντικές, έλαβαν δύο σημαντικές αποφάσεις. Αποφάσεις που μας έφεραν σε αυτήν τη σημερινή κατάσταση και μας υποχρεώνουν να λάβουμε γρήγορα αποφάσεις. Πρώτον, το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισε ότι κράτος όπως ο Ισημερινός ε, που έχει ανάγκη να αναπτύξει την εσωτερική του οικονομία να μειώσει το επίπεδο της ε, φτώχειας και να βελτιώσει το κατακυφερήν εισόδημα των 4.000 δολαρίων έχει προχωρήσει τόσο ώστε θα πρέπει να αποκλειστεί από το σύστημα γενικών προτιμήσεων. Δεύτερον, το Συμβούλιο και αντίστοιχα πλέον ψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτουν ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Κολομβία και το Περού που αρχικά είχαν προβλεφθεί ως περιφερειακές συμφωνίες ώστε να μην τίθεται σε αμφισβήτηση ή ε, να μην τίθεται σε αμφισβήτηση η πορεία ε, του Ισημερινού. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί να κοιτάξει να δουλέψει περισσότερο πάνω στο κράτος αυτό επιλέγει την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τον Ισημερινό. Αυτή την επιλογή έκανε στρατηγικά και ιδιαίτερα στο θέμα του ανταγωνισμού πρέπει να σημειώσουμε ότι και η αλλαγή των παγκόσμιων συνθήκων πλαισίων για ορισμένα σημαντικά ε, εξαγωγικά προϊόντα του Ισημερινού δυσκολεύουν για την κυβέρνηση Κορέα την προσχώρηση στην ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Κολομβίας, που έχουμε με την Κολομβία και το Περού. Αυτό οδηγεί σε δυσκολίες την ε, κυβέρνηση και μπορεί ακόμη να ε, την θέσει σε κίνδυνο, την κυβέρνηση του σημερινού. Αυτό θέλουμε. Έτσι λοιπόν, πρέπει να συνεχίσει το σύστημα των προτιμήσεων μέχρι ότι μπορεί να τεθεί σε, εφαρμογή το, η Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου. Χρειάζεται να δώσουμε αυτή τη γέφυρα μετάβασης για το λαό του Ισημερινού. Ξέρω ότι εσείς κυρία Επίτροπε με τα τωρινά σας καθήκοντα ήδη γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης για τον Ισημερινό. Αποφασίσατε δηλαδή να έχετε τη δυνατότητα ανα πάσα στιγμή να πιέσετε πολιτικά τη χώρα. Ανα πάσα στιγμή που ο Ισημερινός θα μπορούσε ενδεχομένω να εισαγάγει μέτρα ε, που θα ενοχλούσαν την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Οι δικές μου προτάσεις και οι τροπολογίες με τις οποίες προσπαθώ να υποβαθμίσω την ε, κρίση δυστυχώς δεν έχουν εξασφαλίσει πλειονοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Η κεντροδεξιά πλειονοψηφία αποφασίζει να παραιτηθεί από τα δικαιώματα και τις προνομίες του Κοινοβουλίου και να επιτρέψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάσα στιγμή να διατυπώνει την αρνησή κυρία τη, παρά το γεγονό ότι η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου η οποία μελέτησε τη διαδικασία της ε, κατεξοδότησης πράξης και την προτείνει ως απαραίτητη, ε, τίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ελπίζω ότι αυτό το λάθος δεν θα αποτελέσει προηγούμενο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με όλα αυτά απευθύνω για μια τελευταία φορά έκκληση να υποστηρίξετε και να εγκρίνετε τον καρονισμό για να βοηθήσετε τον λαό του σημερινού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόλτς. Δουλεύει τώρα το μικροφωνό μου και δίνω το λόγο στην κυρία Μάλστρομ, την Επίτροπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σημερινού. Μερικά χρόνια μετά την αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις το 2009 επανήλθε σε αυτές και θέλει ο σημερινός να, ε, να ξαναενταχθεί ε, και πάλι στις ε, διεθνείς αυτές διαπραγματεύσεις για να δημιουργηθεί αυτή η ζώνη ε, των συναλλαγών και μάλιστα συναντήθηκα και με τον Υπουργό πριν από 10 μέρες περίπου για να μπει ο Ισημερινός στην ε, συμφωνία, για να ενταχθεί στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, χωρών ε, βολιβίας ε, των χωρών των Άνδεων. Πρέπει να σας πω πως με αυτή την προοπτική θα πρέπει να θεωρήσουμε πως ο κανονισμός αποτελεί και μια, ένα πολύ σημαντικό συνοδευτικό στοιχείο της ε, ίδιας της συμφωνίας. Να είμαστε σίγουροι λοιπόν πως για το προτιμησιακό καθεστώς, εάν προσχωρήσει σήμερα ή σημερινός, να μην υπάρχει καμία αλλαγή. Θα ήθελα λοιπόν να σας παροτρύνω να επεκτείνουμε αυτές τις προτιμήσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στις εξαγωγές της χώρας αυτής. Ο σημερινός ξέρετε πως θα είναι από το γενικευμένο σύστημα ε, συν ε, θα το ξεπεράσει σήμερα και πρέπει να σα πω πω το 60% των εξαγών τη χώρα αυτή εμπίπτουν σε αυτό το καθιστό. Έτσι ώστε να γεφυρώσουμε λοιπόν αυτό το χάσμα μέχρι η συμφωνία να ισχύσει πλήρω και να υπάρχει η βεβαιότητα στους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και κυρίω σε επίπεδο εργαζομένων στο Εκουαντορ. Αν λοιπόν καταφέρουμε ε, να το γεφυρώσουμε έχει καλά. Διαφορετικά ε, θα μειωθεί ε, η εμπορική σχέση μεταξύ των χωρών μας θα αυξηθούν οι δασμοί για τον Ισημερινό και καταλαβαίνετε πως αυτό θα οδηγήσει ε, και σε μία μείωση των εμπορικών μας σχέσεων και η δασμοί θα αυξηθούν κατά 20% για τον τόνο και τις γαρίδες και κατά 15% για όλες τις εξαγωγές του Ισημερινού προς τη χώρα μας. Ξέρω πως οι ευρωβουλευτές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη συμφωνία αυτή και κυρίως στην ε, ρήτρα για την ε, ε, συμμόρφωση με τις διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα από πλευρά σημερινού, όπως επίσης και για τη ρήτρα αναστολής. Είναι σημαντικό λοιπόν, το έθιξα και με τον ε, Υπουργό, με τον οποίο συναντήθηκα την περασμένη εβδομάδα, και να είστε σίγουροι πως εμείς θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση και θα σας τηρούμε ενήμερους για το πώς αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται οι διατάξεις. Όποτε χρειαστεί θα έρθουμε εδώ για να σας δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται και να εξασφαλίσουμε διαφάνεια στην εφαρμογή του κανονισμού, όπως επίσης και να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές τις οποίες έχουμε ε, αναπτύξει στα πλαίσια άλλων συμφωνιών ε, ε, γενικών προτιμήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρώτος ομιλητής από τις πολιτικές ομάδες, από το ΕΛΚ, έχουμε τον κύριο Φίσα Σαϊσέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Επίτροπο και την κυρία Πρόεδρο. Τον Ιούλιο τελείωσαν οι διαπραγματεύσει για την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Σημερινού. Το ΕΛΚ πιστεύει πω η συμφωνία αυτή θα είναι πάρα πολύ ευνοϊκή και για τα δύο μέρη, παρόλο που θα καθυστερήσει δύο χρόνια περίπου να τεθεί σε ισχύ. Από τον Ιανουάριο θα πάψει ε, ο Ισημερινός να χρησιμοποιεί τα πλονεκτήματα που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 προσφέρει η Συμφωνία Γενικευμένων Προτιμήσεων ΣΥΝ. Η πρόταση λοιπόν κανονισμού προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα του χάσματος ε, μεταξύ της θέσης σε ισχύ και της λήξης του συστήματος και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ εμείς ε, υπερψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία χωρίς καμία τροπολογία αυτή την πρόταση για να μην παρατείνουμε χωρίς λόγο αυτές τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων. Η έγκριση αυτού του κανονισμού θα επιτρέψει και η εξαγωγή αλλά και η εισαγωγή να συνεχίσει να εμπορεύονται με φυσιολογικούς ρυθμούς χωρίς να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη αύξηση των δασμών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, ε, βλάβες που δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπεράσουμε και ε, στην Ευρώπη αλλά και στον Ισημερινό. Και μιλώ και για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Ισημερινό. Θα πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε αυτόν τον κανονισμό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Δεν θα ήθελα να κλείσω χωρίς να καλωσορίσω τον Διεθνή Σημερινό στις συμφωνίες αυτές, στις διεθνείς συμφωνίες ε, ελεύθερου εμπορίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος για τους οσυλλοδημοκράτες, ο κύριος David Martin. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον εισηγητή για τις προσπάθειες που έκανε. Εμείς στηρίξαμε στην Επιτροπή της τροπολογίας τους και Νομίζω πως ε, καλά έκανε και δεν τις επαναφέρει στην Ολομέλεια για να μην καθυστερούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισημερινού στις εξαγωγές. του οποιαδήποτε παρακόλληση του εμπορίου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία του Ισημερινού με πιθανότητα το αποτέλεσμα οι να ψάξουν για άλλες αγορές με ευκολότερη πρόσβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ε, πρόταση αυτή που γεφυροποιεί το κενό που δημιουργήθηκε θα συνεχίσουν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισημερινού και θα συνεχίσουν και τα δύο μέρη να ευνοούνται από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Χαίρομαι γιατί μέσω αυτής της ε, ρήτρα αμοιβαιότητας τα ίδια πλεονεκτήματα θα προσφερθούν και στους Ευρωπαίους εξαγωγείς προς τον Ισημερινό και χαίρομαι Επίσης για τις ρήτρες δρασφάλισης που υπάρχουν στη Συμφωνία για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Νομίζω πως είναι μια καλή συμφωνία για όλους. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εσάς την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τον εισηγητή. Ε, Mr. ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Ο κύριος Ραμόν Τρεμόσα Ιμπαρσέλς έχει το λόγο για 1,5 λεπτό από τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί Επίτροποι, πε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συζήτηση. Χαιρετίζω την ε, συζήτηση και μετά την θετική ψήφο στην ΙΝΤΑ έπρεπε το θέμα αυτό να εγκριθεί από την Ολομέλεια πριν από το τέλος του έτους γιατί πολλές οικονομικές συμβάσεις των Ισημερινών θα πρέπει να τύχουν διαπραγμάτευσης τώρα πριν από του χρόνου. Νομίζω ότι οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου περισσότερο από το δημόσιο χρέος μπορούν να, να βοηθήσουν την Ευρώπη να φτάσει προς την ανάπτυξη. Υποστηρίζω τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανοίξει νέες αγορές και να μειώσει τους δασμούς. Στην Ίντα εμείς καταψηφίσαμε τις τροπολογίες του εισηγητή διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Υποστηρίζω την, το προτιμησιακό καθεστώς των ε, αγαθών από τον ε, Ισημερινό πριν τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και θεωρούμε ότι θα ανοίξει ο Ισημερινός ε, τις, επιχειρήσεις, τις αγορές συγγνώμη, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επίσης η στάση της Ρωσίας θα πρέπει να μας οδηγήσει να βρούμε νέες αγορές στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Ευχαριστούμε κύριε Τρεμόσα. Η κυρία Σκακέλερ, πράσινη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ τον εισηγητή για την ίδια την έκθεση, μάλλον για την ουσία της, όμως δεν είμαι τόσο ικανοποιημένη, γιατί όπως ε, είχε επισημάνει και ο εισηγητής κύριος Σόλτς, δείχνει αυτή η υπόθεση το πώς ε, δεν βοηθάει το εμπόριο την ανάπτυξη. Δηλαδή, είχαμε ένα σύστημα που υποχρέωνε τις αναπτυσσόμενες χώρες να κάνει μια επιλογή εάν θέλει να παραιτηθεί από την προτιμησιακή μεταχείριση για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά ή αν θέλει να υπογράψει σύμβαση ελευθέρου εμπορίου. Κάτι το οποίο όμως δεν θα πρέπει να γίνεται και έξω από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και με τον εκβιασμό και την υπονόμευση των δικαιωμάτων του κράτους. Αυτό συμβαίνει εδώ με τον σημερινό. Ή χάνει την προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά ή ακολουθεί την πορεία του Περού και της Κολομβίας. Και γι' αυτό κύριε Επίτροπε σας καλούμε εδώ να ξανααναλογιστείτε την ε, πρόσβαση στο εμπόριο και την ανάπτυξη ως μέσα, γιατί το εμπόριο αυτή τη στιγμή ε, υπονομεύει την ανάπτυξη. Πρέπει να κάνουμε μια πιο σοβαρή μελέτη της υπόθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ατόντο έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σόλτς γιατί φάνηκε πραγματιστής. Σημεριστήκαμε τη στάση του ως προς τις τροπολογίες και θεωρώ ότι υπάρχει ευεργέτημα για τον σημερινό βάση αυτού του κανονισμού. Θα ήθελα να σας πω ότι ίσως η Ευρώπη λαμβάνει μία σημαντική απόφαση και για την ίδια. Γιατί ως πρόεδρος της Eurolat θα ήθελα να σας πω ότι όλο ένα και περισσότερο από τη Λατινική Αμερική υπάρχει στάση να κοιτάν προς τον ειρηνικό και όχι προς την Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε την εμπορική μας δραστηριότητα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει μεγάλη ευθύνη διότι εμείς προωθούμε τη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική αλλά δυστυχώς μας υποκαθιστά η Κίνα και η Ρωσία στη Λατινική Αμερική. Γι' αυτό θα πρέπει να ευεργετηθούμε από αυτή τη συμφωνία, γιατί έχει μεγάλη πολιτική σημασία ως προς τις σχέσεις με την Λατινική Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Κέρθεν Ντάρλιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο η θα ε, συμμετάσχει στην ε, Συμμαχία Εμπορίου με την Κολομβία και το Περού. Και θα ήθελα ο κανονισμός αυτός να διασφαλίσει ώστε το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισημερινού να μην διαταραχθεί πριν ψηφιστεί αυτή η συμφωνία. Και θα ήθελα να δείξω και ένα άλλο σημείο. Πριν από δύο χρόνια εγκρίναμε ένα ψήφισμα ζητώντας από τις χώρες των Άνδεων και ιδιαίτερα τότε την Κολομβία και το Περού να δεχτούν οδικούς χάρτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιβαλλοντικές συμφωνίες. Θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο για τον Ισημερινό, διότι οι εμπορικές μας συμφωνίες δεν, αφοράν, δεν αφορούν αποκλειστικά το δασμολόγιο. Θέλουμε όμως να βελτιώσουμε την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό θα ήθελα να προωθηθεί ο δικός χάρτης και με τον Ισημερινό. Στο ε, το λόγο έχει ο κύριος Ντάνιελ Κασπάρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε συνάδελφοι. Είμαι ευγνώμων στον εισηγητή γιατί με τον τρόπο του μας επιτρέπει να, να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση για το σημερινό των δασμολογικών, των εμπορικών προτιμήσεων για να προχωρήσει μετά στην εμπορική συμφωνία. Θα ήταν βέβαια γελίο να τιμωρείται πρώτα μια χώρα η οποία συνάπτει μαζί μας συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την απώλεια των προτιμήσεων και να υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες που ανέφερε και η κυρία Κέλλερ. Και γι' αυτό απευθύνω έκλειση στην ομάδα σας. Εάν θέλουμε την ανάπτυξη, εάν δεν θέλουμε εμείς να κυδαιμονεύουμε τους πολίτες στη χώρα αυτή, αλλά να στηρίξουμε τη δημοκρατική κυβέρνηση της χώρας που θέλει να βοηθήσει, να προωθήσει την ανάπτυξη της χώρας, πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Δημοκρατία είναι αποφάσεις είναι η πλειονοψηφία αποφασίζει και η μειονοψηφία πρέπει να τη δέχεται την απόφαση της. Χαίρομαι λοιπόν που θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε ακόμη αυτήν την εβδομάδα και ιδιαίτερα για τα πλέον εκτήματα που θα προσφέρει αυτή η συμφωνία για όλους τους πολίτες στην Κολομβία, το Περού αλλά και τον Ισημερινό. Σας ευχαριστώ κύριε Κασπάρη. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Κύριε Μάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που έγινε. Μέσω της υιοθέτηση αυτού του κανονισμού οι εξαγωγές ε, δεν θα επηρεαστούν μέχρι να μπει σε ισχύ η συμφωνία. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό ενδιάμεσο βήμα που στέλνει ένα πολύ στεναρό μήνυμα και σε επιχειρήσεις που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα στις εξαγωγικέ δραστηριότητες αλλά και ένα πολιτικό μήνυμα στον Ισημερινό η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει στενότερες σχέσεις και θα προχωρήσει γρήγορα προς τη θέση σε ισχύ της ίδια τη συμφωνίας και θα επιτρέψει στον Ισημερινό να διαφοροποιήσει την οικονομία του περισσότερο και να εξαλείψει σε μεγαλύτερο βαθμό τη φτώχεια. Αυτή τη στιγμή προχωράμε προς τη θέσει σε ισχύ τη συμφωνία. Ελπίζω πως το πρωτόκολλο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συγκατάθεση κάπου στα μέσα τη επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή για τα όσα έκανε και για το ότι τόσο γρήγορα διεκπαιρέωσε αυτό το φάκελο. Η καλή εφαρμογή αυτού θα δώσει μια απόκριση στις ανησυχίες που κάποιοι είχαν σήμερα ε, εκφράσει. Κυρία Κέλλερ, σύμφωνα μαζί σας, η το εμπόριο είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να βοηθήσει στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να αναπτυχθούν και να μπουν στην εμπορική μας κοινωνία. Είναι σαφέστατα κομμάτι των προτεραιοτήτων μου αυτό και ξέρετε πως στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάσαμε και μια νέα εμπορική στρατηγική όπου το στοιχείο αυτό και πάλι θα ε, στηριχθεί από εμάς. Ε, το συζητάμε και στις συναντήσεις μεταξύ επιτρόπων, αλλά θα περνάνε τα θέματα αυτά και από εσάς. Μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς σίγουρα θα έχετε νέα. Και θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω τους Ευρωβουλευτές για την καλή συνεργασία μέχρι σήμερα και με χαρά περιμένω ε, και προσμένω στην συνεργασία μας και το επόμενο έτος. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση δεν έχει κλείσει ακόμα γιατί έχουμε ακόμα ε, τον εισηγητή, στον οποίο δίνω τώρα το λόγο. Κύριο Σέλμουντ Σόλτς. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είμαι τι άλλο κατέστησα σαφές ότι υπάρχει βούληση ισχυρή για καλές σχέσεις ε, με το Ευρω... μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ισημερινού και πρέπει να πούμε ότι δεν αρκεί πάντοτε το να λαμβάνονται δημοκρατικά οι αποφάσεις. Μπορεί να είναι καλές οι εμπορικές σχέσεις, αλλά πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ισότιμο. Τον επόμενο μήνα θα έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης να, να εξετάσουμε τη συμφωνία, ιδιαίτερα τις συνέπειές τους προς την απασχόληση, την ποιότητα ζωής του πληθυσμού, το περιβάλλον, αλλά και εν γέννη τη σταθερότητα και τη δημιουργία συνθήκων για ολόκληρη την περιοχή, κύριε Κασμάρη. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ την Επιτροπή να σταματήσει να παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική κατάσταση της ε, χώρας και της περιφέρειας αυτής με κυβερνήσεις που έχουν αποφασίσει να αλλάξουν πορεία και να εγκαταλείψουν τα νεοφιλελεύθερα, πιστεύω, για να δώσουν μια νέα ελπίδα στη χώρα τους. Εγώ ως εισηγητής θα παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή εάν η Επιτροπή έστω και έμεσα κοιτάξει να ζητήσει από τον Ισημερινό τροποποίηση μέχρι και του συντάγματό του για να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις δημόσιες προμήθειες και υπηρεσίες. Και επίσης θα ήθελα να ζητήσω έναν οδικό χάρτη, ένα φύλλο πορεία, όπω άλλωστε υπογράμμισα και νωρίτερα, που θα καταγράφει την πορεία για την πρόσβαση στη Συμφωνία Εμπορικών Συναλλαγών με την Κολομβία και το Περού, χωρίς όμως αυτό να επιδεινώνει τις συνθήκες για τον Ισημερινό. Ορόσημα δηλαδή για την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή κύριο Σόλτς και επίσης θα ήθελα και εγώ να εκφράσω ευχές για καλά Χριστούγεννα και ελπίζω να μπορέσετε να ξεκουραστείτε στις διακοπές κυρία Επίτροπε και εύχομαι κάθε καλό για τον